δάφυλλο και όχι κόκκινο οπότε θα μας εξηγήσετε γιατί. Σχετικά με το ε, εσωτερικό κανονισμό οι φιλελεύθεροι ε, έχουν, ε, ο κύριος Παπαστάμκος μάλλον έχει ζητήσει το λόγο. Προς εμάς και δημών προς το σώμα όπως προταχθεί για ευεξήγητους λόγους η ψήφιση της έκθεσης του κυρίου συναδέλφου κυρίου κρίς Ντέιβις. Σας ευχαριστώ. Είναι κάποιος υπέρ αυτής της προτάσεως. Κάποιος ο οποίος είναι αντίθετος. Ο κύριος Λάινεν. Ε, ε, πρόεδρε, είμαι αντίθετος. Ε, το ΕΛΚ μας εκπλήσει και έχει συζητηθεί η πρόταση αυτή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχει γίνει καλή συνεργασία με την Επιτροπή Γεωργία. Συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Βιομηχανία πρέπει να γνωρίζει πόσο θα κινηθούμε για την κλιματολογική προστασία και θα ήμουν υπέρ του να ψηφίσουμε σήμερα. Ε, Η παράκλησή μου δεν αφορούσε να μην ψηφιστεί σήμερα, να προηγηθεί στη διαδικασία τη ψηφοφορία, Να ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση του Chris Davis. Υπήρξε ένα, ε, υπήρξε μια παρανόηση. Ε, ναι, ε, ίσως η μετάδοση δεν ήταν τελείως ε, ορθή. Άρα ο κύριος Παπαστάμκος ε, ζητά να ψηφιστεί πρώτα η έκθεση Davis. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ του να, υπερψηφι... να ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση Davis. Κατά. Ωραία. Αυτή είναι, όντως είναι πλειοψηφία. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Τώρα θα ψηφίσουμε ε, για ε, να ξεκινήσουμε με την έκθεση Davis. Με συγχωρείτε πρέπει να τακτοποιήσω τα έγγραφά μου λέει ο πρόεδρος και ξεκινάμε με την έκθεση Davis ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 ξεκινάμε με την πρώτη τροπολογία 27 ψηφίσατε όλοι λίγοι Απερίφθη. Ε, τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Ξεκινούμε με το πρώτο τμήμα. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απερίφθη. Δεύτερο τμήμα. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι. Λίγοι. Απερίφθη. Ερχόμαστε τώρα στο αρχικό κείμενο της παραγράφου 2, πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποδεκτή. Ε, και ονοματιστική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα, η οποία ξεκινά ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απερίφθη. Τρίτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απερίφθη. Σωστά το είδαμε. Το τέταρτο με, ε, τμήμα ονομαστικά ξεκινά. Ψηφίσατε. Λίγοι. Απερίφθη. Ερχόμαστε τώρα στο αρχικό κείμενο της παραγράφου 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά. Ψηφίσατε. Λίγοι. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Μάλλον παράγραφος 6, δεύτερη τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απερίφθη. Παράγραφος 15. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Παράγραφος 23 στο αρχικό κείμενο. Ε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 5 ονομαστική πληροφορία για το πρώτο τμήμα. Ξεκινά. Ψηφίσατε. Λίγοι. ενεκρίθη. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 5 ξεκινά ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε, λίγοι. Ενεκρίθη. Οπότε αλλάζει το αρχικό κείμενο και έχουμε την τροπολογία 6 ε, όλοι ηλεκτρονικά υπέρ ε, ψηφίσατε Ξαναρωτάω, ψηφίσατε. Λίγοι. Ενεκρίθη. Το αρχικό κείμενο τώρα καταργείται. Και ερχόμαστε στην παράγραφο 24 με ονομαστική ψηφοφορία που ε, ξεκινά ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Λίγοι. εγκρίθηκε. Τροπολογία 7, δι, ε, ονομαστικά, ξεκινά ηλεκτρονικά, ψηφίσατε, λίγοι, ενεκρίθη. Τροπολογία 8, ονομαστική ψηφοφορία, ξεκινά. Ψηφίσατε, λίγοι. ενεκρίθη. Ερχόμαστε στην τροπολογία 9β, ονομαστική ψηφοφορία, ξεκινά ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Λίγοι. Ενεκρίθη. Τώρα τροπολογία 14 ονομαστικά ηλεκτρονικά ξεκινά Ψηφίσατε λίγοι. Απερίφθη. Τροπολογία 10 ε, ονομαστικά. Ψηφίσατε. Λίγοι. Ενεκρίθη. Το αρχικό κείμενο της, ε, του παραγράφου 27 υπέρ κατά αποχές απερίφθη παράγραφος 28 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη προφανώς απερίφθη και ερχόμαστε στην παράγραφο 31 όπου υπάρχουν ε, τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος ξεκινά ψηφίσατε λίγοι ενεκρίθη δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά ψηφίσατε λίγοι απερίφθη Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. Ελέγχουμε και πάλι. Ξεκινά. Ψηφίσατε. Λίγοι. Απερίφθη. Τώρα το αρχικό κείμενο παραγράφου 42 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Με συγχωρείτε, κάποιο λάθος έκανα διότι ε, πρέπει καταρχήν να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο της παραγράφου 38 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Παράγραφος 38, αρχικό κείμενο, ξεκινά, λίγη. Παραμένει. Εφόσον υπάρχει ισοψηφία παραμένει το αρχικό κείμενο. Το παράγραφος 42. Πρώτο τμήμα διανατάσεως χειρών υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ξεκινά. Ψηφίσατε, λίγοι. Ενεκρίθη. Παράγραφο 44 χωριστά. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές ενεκρίθη δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη παράγραφο 45 καταρχήν η τροπολογία 12 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά ψηφίσατε όλοι λίγοι ενεκρίθη ε, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απερίφθη αρχικό κείμενο σε ονομαστική ψηφοφορία ξεκινά ηλεκτρονικά ψηφίσατε λίγοι ενεκρίθη Τροπολογία 20 Δέλτα υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 21 ονομαστική ψηφοφορία ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Απερίφ, ε, κλείνει. Απερίφθη το κείμενο της παραγράφου 22 ω ε, η ονομαστική ψηφοφορία λίγη απερίφθη τροπολογία 4 οπότε ε, ε, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απερίφθη Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο. Με ονομαστική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα ξεκινά. Ψηφίσατε λίγοι. Ενεκρίθη το δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινά. Ψηφίσατε. Λίγοι. Ενεκρίθη. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά ενεκρίθη δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίσατε όλοι λίγοι απερίφθη τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Παράγραφος 79 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά. Αποχές ενεκρίθη. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Αποχές ενεκρίθη. Παράγραφος 83 του αρχικού κειμένου υπέρ σε δύο τμήματα. Κατά. Αποχές ενεκρίθη. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Αποχές ενεκρίθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος εφόσον το επιθυμείτε ξεκινά για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 83. Ψηφίσατε. Λίγοι. Απερίφθη. Παράγραφος 88. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές Ενεκρίθη Δεύτερο τμήμα υπέρ Κατά Αποχές Ενεκρίθη Ξεκινάει η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 88. Λίγη. Ενεκρίθη. Ε, τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο του 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε στο αρχικό κείμενο της παραγράφου 96 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά. Αποχές. Ενεκρίθη. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινά. Ψηφίσατε. Λίγοι. Παραμένει το αρχικό κείμενο. Ε, ψηφίζουμε την τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές Μου φαίνεται ότι ενεκρίθη. Ενεκρίθη. Αρχικό κείμενο. Άρα, τροπολογία, ε, παράγραφος 15, ε, τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Αλλά αν δεν σηκώνετε το χέρι σας δεν σας βλέπω. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ενεκρίθη αρχικό κείμενο της παραγράφου 107 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αρχικό κείμενο της παραγράφου 110 υπέρ κατά αποχές μου φαίνεται ότι ενεκρίθη ηλεκτρονικός έλεγχος Ξεκινά ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απερίφθη. Είχατε δίκιο. Ερχόμαστε τώρα στην παράγραφα 115 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ε, το δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία ξεκινά ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Λίγοι. Απερίφθη. Πα... Τροπολογία 26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απερίφθη. Το εκτιμώντας ε, β σε δύο τμήματα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα ε, ονομαστικά ξεκινά ηλεκτρονικά η ψηφοφορία ψηφίσατε λίγοι απερίφθη τώρα έχουμε το συνολικό κείμενο ηλεκτρονικά ε, ξεκινά για ονομαστική ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Ενεκρίθη. Τώρα όσον αφορά τι τόπο που γεννούν διακρίσεις και κυβερνητικέ αντιδράσεις ε, θα ψηφίσουμε συλλογικά όλες τις προτάσεις. Πρώτη τροπολογία ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το Έμ στο αρχικό κείμενο. Ψηφίσατε. Εγκρίθηκε. Συνολική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε στα ψηφίσματα σχετικά με τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά αποχές θα έλεγα ότι υπήρξε απεργία ψηφίσματος ε, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απερίφθη Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ούτως ή άλλως, αφού δεν σηκώνετε τα χέρια σας, καλύτερα ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγοι. Ενεκρίθη. Πολύ ωραία. Τροπολογία 5. Ε, υπάρχει μία προφορική τροπολογία του κυρίου Σαλαφράνκα. Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να υπάρχει μέγιστη δυνατή συνένεση, διότι θεωρούμε ότι το ψήφισμα αυτό θα πρέπει να έχει μεγάλη στήριξη από την Ολομέλεια, προτείνουμε μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία 5. Συμφωνούν και ο κύριο Φερχόψτα και ο κύριο Βόμποντα και οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε και θα θέλαμε να προσθέσουμε τον όρο introduction and strengthening and implementation και να αντικαταστήσουμε το condense από το regrets. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι κάποιος ενάντιος σε αυτό. Όχι. Οπότε με την προφορική τροπολογία του κυρίου Σαλαφράνκα ψηφίζουμε την τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και ε, τα πίπτη το 14, τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 15 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται υπέρ 11 υπέρ κατά αποχές πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος Ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απερίφθη. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 12 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 16 πρέπει να ψηφιστεί ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το 12 απεσήφθη ε, το 2 απεσήφθη 3 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 8 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 1 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη αποσύρεται το 13 το 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 9 υπέρ κατά αποχές εν, ε, απερίφθη ε, το ψηφίζουμε το συνολικό κείμενο. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε ε, ε, στο ψήφισμα για το Καζακστάν. Η κυρία Γιακονσάρη. Έχω πολύ καλά νέα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας οι αρχές του Καζακστάν απελευθέρωσαν πολιτικούς ε, κρατομένους. Ε, την κυρία Σοκόλοβα συγκεκριμένα και σήμερα τον αρχή συντάκτη Ιγκορ Βινιάρσκι. Ευχαριστώ κυρία Γιακονσάρη για τα καλά νέα. Η τροπολογία 7 ξεκινά ονομαστικά. Ψηφίσατε λίγοι. Απερίφθη. Παράγραφος 3 σε 2 τμήματα για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάει. Ψηφίσατε. Λίγοι. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ενεκρίθη. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη το αρχικό κείμενο της παραγράφου 10 σε 3 τμήματα υπέρ κατά αποχές για το πρώτο τμήμα ενεκρίθη παρακαλώ να σηκώνετε κυρίες και κύριοι τα χέρια σας διαφορετικά μαντεύω και δεν μιλάμε για μαντίες εδώ τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 12 του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη παράγραφος 13 πρώτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά ψηφίσατε λίγοι ενεκρίθη το 2 καταπίπτει 3 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη η τροπολογία 4 με ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινά ψηφίσατε λίγοι απερίφθη ερχόμαστε στο αρχικό κείμενο ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ενεκρίνεται τώρα τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη και ψηφίζουμε το συνολικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. Τώρα έχουμε την ψηφοφορία για την κατάσταση στην Ιγυρία. Έχουμε ε, μία, ένα κοινό ψήφισμα από έξι πολιτικές ομονόνδες που ψηφίζεται υπέρ κατά αποχές νεκρήθη το ψήφισμα. Τώρα ερχόμαστε στην κατάσταση Λευκορωσία όπου ο συνάδελφος Βιγγένιν έχει ζητήσει το λόγο. Χθε πρόεδρε είχαμε μια αναλυτική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήταν σαφές το μήνυμα Υπάρχει μια κοινή πρόταση ψηφίσματος, ένα σχέδιο ψηφίσματος πολύ ξεκάθαρο. Είναι ε, συσπηρωμένο το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει προς ε, την ε, κοινωνία της Λευκορωσίας, την ηγεσία της Λευκορωσίας αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη θα έλεγα, ε, για δύο λόγους. Ε, για να δοθεί χρόνος ε, στις αρχές να ανταποκριθούν, να αντιδράσουν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται και για να μπορούμε να τροποποιήσουμε το ψήφισμα τις τελευταίες εξελίξεις που αναμένουμε να αναβληθεί ψηφοφορία για την μηνυλομέλεια των Βρυξελών. Ευχαριστώ κύριε Βιγγένιν. Κάποιο στηρίζει την πρόταση Βιγγένιν, κάποιο είναι αντίθετος στην πρόταση Βιγγένιν. Κύριε Βουλευτά. Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω πολύ καλά τον κύριο Βικένιν. Πράγματι συζητήθηκε διαμακρών το θέμα. Ο κύριος Λουκασέγκο προχώρησε σε κάποιες ε, χειρονομίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσει η γλώσσα της διπλωματίας και όχι η επιθετικότητα. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα για να δείξουμε και στο Λουκασέγκο ότι είμαστε ενωμένοι. Ας ψηφίσουμε σύμφωνα με το άρθρο 177 στην επό... να ε, γίνει ψηφοφορία στην επόμενη ε, ποιος είναι υπέρ της προτάσεως Βιγγένιν. Κατά. Αποχές έγινε αποδεκτή η ε, απόφαση να μεταφερθεί η ψηφοφορία αυτή στην ε, μήνυ Ολομέλεια των Βρυξελών. Ερχόμαστε τώρα στο έκτο Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό και ζητώ να ψηφίσουμε τη, ονομαστικά την τροπολογία 2. Ξεκινά, λίγη. Απερίφθη. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ξεκινά ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισε, ε, ψήφισαν όλοι. Ενεκρίθη. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη Τέσσερα. υπέρ κατά αποχές Πέντε. υπέρ κατά έλεγχος Ξεκινάει ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε. Λίγοι. Ενεκρίθη. Παράγραφος 8 του αρχικού κειμένου. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές ενεκρίθη. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές ενεκρίθη. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές και 7 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος πρέπει να, πάλι να ελέγξουμε ε, λυπούμε ψηφίσατε ηλεκτρονικά δηλαδή όσοι δεν έφυγαν για να πάνε στο φόρουμ για το νερό απερίφθη η τροπολογία συνολικό κείμενο ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι να γυρίσετε καλά στο σπίτι σας και καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίε e, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου.